και κύριοι συνάδελφοι, στην ημερήσια διάταξη είναι η προσωρινή έκθεση του κυρίου Γιακολίνο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλέσω τον εισηγητή να πάρει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εδώ και πολλά χρόνια συζητάμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να επικροτήσουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θέλησε να αποστείλει ένα στεναρό μήνυμα για τη δημιουργία ενός κοινού χώρου ποινική δικαιοσύνης με τη δημοσίευση ενός νομοθετικού πακέτου το οποίο περιλαμβάνει τη Eurojust, την Ευρωπαϊκή ε, Εισαγγελία και φυσικά θέλει να αναθεωρήσει και την Όλαφ την υπηρεσία καταπολέμησης απάτης. Θα πρέπει βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι η αδιάκοπη ε, δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εντός της Επιτροπής ΚΡΙΜ, στην οποία εγώ ήμουν ο μόνος εισηγητής, ε, να καθορίσουμε κάποιες προτεραιότητες ε, και ένα χρονοδιάγραμμα με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ε, και ένα χρονικό ορίζοντα ε, μεταξύ του 2014 και του 2019 για την καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων και μέσω ενός οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα μπορεί να διώκει αυτά τα εγκλήματα με συγκεκριμένη αναφορά και συγκεκριμένη μνήα ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταπολέμηση της κοινοτικής απάτης μέσω ενισχυμένης ε, δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Ε, πόροι οι οποίοι ε, χάνονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο που χάνονται από την UEFA, από την πολιτιστική συνεισφορά, από τα όσα θα μπορούν να δοθούν σε πάρα πολλά ταλέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά δίνονται για ξέπλυμα χρήματος, για διαφθορά και πολλά άλλα. Κυρία Ρέντινγκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δρά ε, με ευέλικτο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν θα πρέπει να συνεργάζεται με την Eurojust και με την Όλαφ για την κατεπολέμηση της απάτης. Ε, οι σκιώδεις εισηγητές ε, και οι σύμβουλοι μας επέτρεψαν μέσω της συνεργασίας τους να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Υπάρχουν ε, κάποια μέτρα για τους ε, ανθρώπους οι οποίοι είναι αντικείμενο έρευνας. Έχουμε διερευνήσει και κάποια συγκεκριμένα θέματα για τα καθήκοντα της εισαγγελίας και έχουμε εκφράσει και την άποψή μας όσον αφορά τα μέτρα και τις δυνατότητες έρευνες και ανάκρισης το κατά πόσον γίνονται παραδεκτές, παραδεκτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Χρειαζόμαστε περισσότερες διαδικαστικές εγγυήσεις ε, χωρίς ταυτόχρονα να αποδυναμώσουμε και το θεσμικό ε, τμήμα του νομοθετικού μέσου. Ε, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αμφισβητήσουμε το έργο των εθνικών δικαστηρίων και θέλουμε να ενισχύσουμε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με κάποια αναφορά ε, για τη δυνατότητα ε, ποινών. Από εδώ και πέρα ο ρόλος είναι στα χέρια του Συμβουλίου. Αύριο ελπίζουμε κυρία Επίτροπε ότι θα εγκρίνουμε αυτή την ενδιάμεση έκθεση η οποία αποτελεί το αυθεντικό ε, στοιχείο της ε, άποψης της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε μια εισαγγελία η οποία να εργάζεται καλά, να χρησιμοποιεί το, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Ευρωπαϊκό Ένταλμα έρευνα στη δυνατότητα δίμευσης ε, και κατάσχεσης περιουσίας και όταν θα μπορέσουμε να έχουμε έναν ενιαίο χώρο ε, ποινική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Σήμερα στην Ολομέλεια ε, καθορίσαμε και κάποιους περιττέρω κανόνες διαφάνειας που θα δώσουν τη δυνατότητα στον Ευρωπαίο Εισαγγελία να εντοπίζει καλύτερα ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές οι οποίες θα μπορέσουν να αποτελέσουν απάτη ίσως ε, σε κοινοτικό επίπεδο ή διαφθορά. Τα όσα έγιναν στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας ε, θα πρέπει να προχωρήσουν ε, διότι είχαμε ενθερετικά στοιχεία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δε και την αρχή της αναλογικότητας και της επικορικότητας και σε θέματα ποινική δικαιοσύνης. Ολοκληρώνω, θεωρώ ότι η αξιοπιστία ε, και η εμπιστοσύνη προς τους Ευρωπαίους πολίτες προκύπτει και μέσω μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ελπίζουμε ότι οι κοινοτικοί πόροι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να είναι ε, στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο και τώρα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Αντιπρόεδρο Βίβιαν Ρέντινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριε βουλευτέ. Επιτρέψατε μου πρώτα πρώτα να σα πω πόσο αισθάνομαι υποχρεωμένοι και ευγνώμη προ το Κοινοβούλιο, προ ε, τον εισηγητή, του σκιώδη εισηγητέ, διότι κάνετε τη φωνή σα να ακουστεί. Ε, σε μια τόσο πρώιμη φάση αυτής της διαδρομής, της διαδικασίας, γιατί αυτό το μήνυμα που στέλνετε είναι ξεκάθαρο για το πόσο σημαντικό και πόσο επίγον είναι το να βρούμε το καλύτερα μέσα για να προστατεύσουμε τον προπολισμό της Ένωσης από τους εγκληματίες. Θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμβάλει επικοδομητικά σε αυτήν την ενδιάμεση εξαίρετη έκθεση. Και ε, ξέρω ότι θα έχουμε την αμέριστη προσοχή σας και συμπαράστασή σα και ότι θα λάβουμε σοβαρά τα όσα έχετε να συστήσετε στα πλαίσια των ε, διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Είναι κοινό το καθήκον μας, είναι καθήκον να πολεμήσουμε την εγκληματικότητα κατά των οικονομικών συμφωνών τη Ένωση. Και οι απάντε στα κρατημέλη επηρεάζουν τον προπολογισμό και οδηγούν σε σημαντικέ απώλειε και ζημίες. Πολλές εκατοντάδες εκατομμύριων χάνονται έτσι κάθε χρόνο. Βέβαια έτσι υπονομεύεται και δυναμητίζεται η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων προς τα θεσμικά τους όργανα και γι' αυτό τον ε, τρόπο πρέπει, γι' αυτό τον λόγο πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και το έγκλημα. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας πρόκειται να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν το έγκλημα. Ο στόχος είναι οι εγκληματίες οι οποίοι παραβλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ε, έχουμε αυτή την πρόταση που πρόκειται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη διατυπώσαμε τον ε, Ιούλιο, ετήσει το Κοινοβουλίο. Και αυτό αποτελεί ε, κάτι από το νέο πλαίσιο το οποίο έχουμε σχεδιάσει. Έχουμε την οδηγία κατά τις απάτες, έχουμε το θέμα των οικονομικών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά έχουμε και την Eurojust. Οπότε θέλουμε έτσι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο και επίσης αποκεντρωμένο τόσο ώστε να μην έχουμε παράλληλες δομές, ε, βαριές ε, και θα πρέπει να ε, ωφεληθούμε από την υπηρεγνωμοσύνη των κρατών μελών από το, την ένωμη τάξη τους να είναι αποτελεσματική αυτή η υπηρεσία του εισαγγελέως. Αυτό είναι μία εκ ε, απαραίτητων συνθηκών εκ των όνους άνευ, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έτσι αυτή την υπηρεσία και όλες αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές που ε, κατοχυρώνονται από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, επί τη βάση της αρχής της δικαίας δίκης και επίσης για τις αρχές της ισότητας των όπλων όπως επίσης από την αρχή του δεδικασμένου. Ναι, μπει Να μην δικάζεται κανεί ή να μην του επιβάλλεται ποινή δύο φορέ για το ίδιο αδίκημα. Επίση, θα πρέπει να θίξουμε και άλλα δύο σημεία τα οποία αναφέρονται στην ενδιάμεση ε, έκθεση αυτή. Τα δικονομικά δικαιώματα και τα ε, ένδικα μέσα. Συμφωνώ για τα δικονομικά, θα πρέπει να τηρηθούν τα ελάχιστα πρότυπα, τα ελάχιστα στάνταρ όσον αφορά την ποινική ε, δικονομία ε, και γενικό την ποινική διαδικασία σε όλα τα μέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, τόσο ώστε να λειτουργεί άρτια αυτή η υπηρεσία του Ευρωπαίου Εισαγγελία. Επομένω, η πρόταση του κανονισμού αυτού πρόκειται να μας δώσει το, την καλύτερη δυνατή προστασία ε, σε σχέση με τους υπόπτους, τους φερομένους ως ένοχους ε, τα δικαιώματά τους, τα οικονομικά. Νομίζω ότι αυτό ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε ε, τις αρμοδιότητες, τις ερευνητικές, ανακριτικές που η υπηρεσία αυτή του Ευρωπαίου Αγγελία μπορεί να ασκήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κλειδί σε αυτή την ε, πρόταση, ούτως ώστε να έχουμε ένα στεγανό σύστημα προτασίας για τα δικαιώματα των υπόπτων, κάτι το οποίο να έχει τις ρίζες του στο κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και στις εθνικές ενόμες τάξεις και το σχέδιο αυτό του κανονισμού ε, αποδίδει ε, δικαιώματα ή αυτούς τους υπόπτους και αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκούνται σύμφωνα με διατάξεις του εθνικού κειμένου, όπως το δικαίωμα της συλλογής και υποβολή ε, αποδεικτικών στοιχείων. Τώρα, να δούμε τι γίνεται, τι προβλέπουν ε, για τα ένδικα μέσα, ε, τι γίνεται, τι μπορούν να κάνουν επίση ω αναπομπή τα εθνικά δικαστήρια, σύμφωνα με αυτή την πρόταση. Έτσι θεωρούμε ότι θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα απονομή τη δικαιοσύνη και ενιαία εφαρμογή του κανονισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω εμείς ε, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για εναλλακτικέ λύσεις ούτως ώστε να διαπραγματευτούμε το Συμβούλιο αυτέ τι άλλε λύσεις και επίσης να έχουμε πιο ενισχυμένο, αναβαθμισμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης, σας ενημερώνω ότι είχαμε μια πολύ επικοδοματική συζήτηση με τους υπουργούς σε σχέση με αυτό το σχέδιο εικονισμού την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη η Ελληνική Προεδρία ε, πάρα πολύ επιδέξια έθεσε τρία ερωτήματα όσον αφορά κάποια, την κατανομή του έργου, τα δικονομικά ε, και επίσης κάποια άλλα διορθωτικά ζητήματα. Και είπαμε ότι οι στόχοι μας ε, συνενούν τη Γενική Συνένεση και θα συνεχίσουμε την πορεία αυτή και σε τεχνικό επίπεδο. Παραμένω πεπισμένοι ότι όσο περισσότερο συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία τα κράτη-μέλη, τόσο καλύτερο, τόσο περισσότερο τόπο θα πιάσουν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Παντού. Και επίση αυτή η πρόσφατη ζήτηση στο Συμβούλιο μου απέδειξε ότι υπάρχει ε, η ευκαιρία τώρα να συνενώσει προσπάθειε πολλών κρατών μελών και νομίζω ότι αυτά είναι καλά μαντάτα. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να έχει ανοιχτή στάση ε, σε σχέση με την διαδικασία που θα ακολουθεί, τις διαπραγματεύσεις, να φτάσουμε σε έναν συμβασμό, να λάβουμε υπόψη ό,τι συστήνει η ενδιάμεση εκθεσή σας και θα προωθήσει αυτό τις επαφές και συζητήσεις. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Μια που δεν έχουμε εδώ τον κύριο Λαμασούρ, θα ήθελα να ζητήσω την κυρία Γκράσλα να πάρει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι κρίμα το ότι δεν είναι εδώ πέρα το Συμβούλιο και είναι ενδεικτικό της διαδικασίας. Υπάρχει ο κίνδυνος ε, να δημιουργήσουμε με αφέλεια μια Ευρωπαϊκή Αρχή η οποία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία θέλουμε και θα προστατεύσει την δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και ειλικρινά απορώ με αυτό το οποίο πρότεινε η Κομισιόν. Οι αδυναμίε παραμένουν και η βασικότερη αδυναμία είναι η αναποτελεσματική δικαιοσύνη σε κάποια, για να μην πω πολλά, κράτη-μέλη. Και δεν κάνει τίποτα η Κομισιόν γι' αυτό, ανταυτού ε, αποφασίζει να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο δεν λειτουργεί. Έχω κάποιες τροπολογίες, ε, τις οποίες θα ήθελα να στηρίξω και αφορούν την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την κατάργηση της ε, ασυλίας ε, των ε, ευρωϊπαλλήλων για να μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή τη δουλειά της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Κυρία Ρέγνερ, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, είπατε τι κοστίζει το να μην έχουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκατοντάδες εκατομμύρια λίγο πολύ ε, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως ε, υπάρχουν πάρα πολλά ε, πάρα πολλέ περιπτώσει οι οποίε ε, μα δείχνουν πω η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποτελεσμα... ένα αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμηση του εγκλήματο ε, και βλέπουμε πω υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τουλάχιστον σε 14 κράτη-μέλη. Επίση δώσαμε ιδιαίτερο βαρό στην σχέση που θα έχει με τον Όλαφ, τη Eurojust και την Europol. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει εδώ πέρα για να έχουμε ένα ενιαίο συνεκτικό πλαίσιο. Οπότε εμείς λέμε ένα σαφές ναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και μια ρεαλιστική ματιά δείχνει πως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ. Πολιτικών ομάδων και πρώτα θέλω να παρακαλέσω την κυρία Χολμάιερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να πάρει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Χαίρομαι για το ότι εκμεταλλεύεται την ευκαιρία η Κομισιόν να καταπολεμήσει το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ε, και στο πλαίσιο της Αρμόδιας Επιτροπής ε, πως ε, πρέπει να υπάρξει κάποια καταπολέμηση της διαφθοράς του οργανωμένου εγκλήματος και βεβαίως της προστασίας των συμφερόντων της κοινότητας. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως αυτό το οποίο λέει η κυρία Γκρέσλε πως δεν υπάρχουν σαφείς οικονομικές και νομικές αρμοδιότητες ακόμα. Βλέπουμε όμως ε, την επίδραση στον προϋπολογισμό της κοινότητας. Δεν μιλάμε για λαθρεμπόρη ναρκωτικών είτε για οποιαδήποτε άλλη εγκληματική δραστηριότητα. Οπότε θα πρέπει νομίζω να ασχοληθούμε με μια αναδιάταξη των σημαντικών ε, τομέων, όπως παραδείγματο χάρη της Eurojust, της Eurojust, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται τίποτα επιπλέον ως μέσο και προσωπικό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είχαμε έναν ε, μικρό αριθμό ατόμων, 190 άτομα τα οποία ασχολούνται με κάποιες χιλιάδες υποθέσεις. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό, πραγματικά πρόκειται για μια υποστελέχωση των υπηρεσιών, το ίδιο και στη Europol. Πώς είπε από σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα δικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας ε, ε, πλήττουν τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Γι' αυτό η ομάδα μου επί της αρχής είναι υπέρ μιας ευρωπαϊκής αγγελίας. Όμως η πρόταση της Κομισιόν ε, όσο έχει αυτή τη είναι προβληματική γιατί αφενός θέλουμε ευρωπαϊκή εισαγγελία με ευρύτατες αρμοδιότητες και αφετέρου δεν έχουμε κάνει τίποτα όσον αφορά κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως εδώ πέρα απαιτούνται και τα δύο και να φέρουμε τους εγκληματίες ενώπιον της δικαιοσύνης αλλά και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Εμείς βεβαίως εδώ πέρα στη διαδικασία αυτή μπορούμε είτε να συμφωνήσουμε είτε να απόρριψουμε οπότε πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα για το που θεωρούμε πως χρειάζεται βελτίωση. Να αναφέρω κάποια βασικά πράγματα. Τα δικονομικά δικαιώματα πρέπει να απτυχθούν και να εναρμονιστούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, ταυτόχρονα χρειάζεται και κάποια νομική αρρωγή για τους ενδιαφερόμενους. Χρειάζεται επίσης ένα σαφής ορισμός για το πότε θα δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή αυτή εισαγγελία και ο κανόνας, οι κανόνες επίσης για το παραδεκτό των αποδεκτικών στοιχείων δεν πρέπει να είναι ο ελάχιστος κοινό παρονομαστής. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, αρχικά θα ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο για την ε, καταπολέμηση των απατών εις βάρος των οικονομικών σφαίρων της κοινότητας. Όμως, εμείς θέλουμε να δούμε και τα αδικήματα αυτά οπωσδήποτε, αλλά ταυτόχρονα με μια ταυτόχρονη βελτίωση των ε, προδιαγραφών ε, ασκήσεως ε, δικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Πολύ Η, συνάδελφο, Βέμπερ από το Άλντε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεισφορά σε αυτή τη σημαντική έκθεση. Καλώς ορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και με πεπισμένη ότι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφεληθεί από μια ευρεία πρόταση που θα σκοπεύει να δημιουργήσει ένα τομέα ποινική δικαιοσύνη ή ε, δημιουργία μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, που θα προστατεύει τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα τη Ένωση είναι απλώ το πρώτο βήμα. Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι το έσχατο, η έσχατη δοκιμή στη βούληση των κρατών μελών να συμμετέχουν σε ένα σχέδιο που θα γίνει ένα βήμα προς τα μπρος στη διαδικασία ε, της, ε, του των, ε, των νομικών μας συστημάτων. Ε, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν δηλώσει τις διστακτικότητά τους ε, να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σχέδιο, αν και είναι αρκετά παλιά η ιδέα και έχει συμπεριληφθεί στη συνθήκη. Ταυτόχρονα αυτή η προσπάθεια θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και τους Ευρωπαίους νομοθέτες, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τους δύο νομοθέτες δηλαδή αν και η νομική βάση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιτρέπει απόφαση του Συμβουλίου με απλή συνένεση του Κοινοβουλίου, εγώ πιστεύω ότι η δημιουργία της Εισαγγελίας μέσω αυτής της διαδικασίας δεν θα πρέπει να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, των ατόμων για το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο έχει νομοθετική εξουσία. Αύριο θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο. Ε, αν δημιουργεί φορείς ε, με λειτουργίες έρευνας, πρέπει να δημιουργήσουμε και το πλαίσιο για να εγγυηθούμε τα δικονομικά δικαιώματα των ατόπων που είναι αντικείμενο έρευνας, ε, σύμφωνα με την δική μας νομοθεσία για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι πεπισμένη ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ελεγγύη θα είναι η αρχές ε, επί των οποίων πρέπει να βασιστούμε αν θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στη δουλειά που ξεκινάμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βέμπερ. Υπάρχει μπλε κάρτα για σας από τον συνάδελφο Ζιόμπρο. Δέχεστε την ερώτηση μάλιστα, κύριε Ζιόμπρο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πιστεύετε ότι θα ήμασταν πιο αποτελεσματικοί αν ε, αποφασίζαμε να αφήσουμε αυτό το έργο στις ε, εθνικές εισαγγελίε αντί να εξοδεύουμε κάθε χρόνο χρήματα για τη δημιουργία ενός νέου γραφειοκρατικού θεσμού που μπορεί και να μην είναι αποτελεσματικός. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα αρμοδιοτήτων ε, και να υπάρχει και σύγκρουση. Κυρία Βέμπερ. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι συζητήσεις ε, έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν Γι' αυτό, σύμφωνα με τη συνθήκη, είναι σήμερα δυνατό να συσταθεί η εισαγγελία. Δεν νομίζω ότι έτσι όπως ε, έχει σχεδιαστεί αυτός ο θεσμός θα είναι γραφειοκρατικός, γιατί πραγματικά θα συνεργάζεται και θα δρά μέσα από τις εισαγγελίες στα κράτη-μέλη. Εγώ απλώς αυτό που θέλω να δω είναι να τεθούν σε εφαρμογή οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ομάδα των Πρασίνων. Thank you, Chair. First of all... Να ευχαριστήσω καταρχήν ε, την εισηγήτρια και τους Κιώδης για το γεγονός πως λάβαμε αυτή την ενδιάμεση έκθεση. Είναι εξαιρετικό το μήνυμα γιατί χρειάζεται τα θέματα αυτά να το προωθήσουμε. Αυτό που δεν με ικανοποιεί είναι ότι δεν είναι εδώ το Συμβούλιο. Άρα λοιπόν ε, τι κάνουμε. Εμείς στο κάτω-κάτω θα κληθούμε στο τέλος να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Και αν δεν είναι εδώ το Συμβούλιο να μας ακούσει σήμερα, τι είδου συγκατάθεση θα δώσουμε. Υπάρχουν κάποιε προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, ότι Εάν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη διασυνοριακή συνεργασία, η οποία είναι όντω απαραίτητη, τότε για να γίνει το Α θα πρέπει να έχουμε Β κοινά πρότυπα και κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο που βρισκόμαστε όλοι μαζί να κάνουμε και να διεκδικήσουμε το δικαίωμα για την ενημέρωση, για την ε, διερμηνία, για την νομική αρρωγή και πρόσβαση σε δικηγόρο, ε, όλα αυτά τα οποία έχουμε συμπεριλάβει. Και μετά έχουμε το επόμενο βήμα. Έχετε δει την οδηγία για την προστασία δεδομένων που ε, έχουμε πάρα πολλούς βουλευτές εδώ που δεν θέλουν να στηρίξουν αυτούς τους κανόνες και τα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το μηδέν και ας οικοδομήσουμε αυτό που χρειάζεται εδώ για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άλμπρεχτ. Μια που αναφερθήκατε την, στην έλλειψη, της, στη μη παρουσία εδώ του Συμβουλίου, θα ήθελα να συστήσω να συζητηθεί το θέμα αυτό με τις πολιτικές ομάδες, γιατί οι πολιτικές ομάδες ε, αποφασίζουν να μυρίσει η διάδειξη σε σχέση και με την παρουσία του Συμβουλίου. Ε, νομίζω ότι από την ΚΟΕ είναι η κυρία Κάρη. Ευχαριστώ πολύ. Έκανα μια πρόταση πως το Κοινοβούλιο θα έπρεπε την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την απορρίψει και θα ήθελα να παρακαλέσω το Συμβούλιο να κάνει το ίδιο. 14 εθνικά κοινοβούλια σε 11 διαφορετικά κράτη-μέλη έχουν σηκώσει κίτρινη κάρτα για την πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα εθνικά κοινοβούλια θεωρούν πω η πρόταση αυτή παραβιάζει την αρχή τη επικουρικότητα και πάει υπερβολικά μακριά. Κάποια κοινοβούλια δεν λένε πω η ε, πρόταση αυτή θα αποτρέψει τα κράτη-μέλη από το να αποφασίζουν τα ίδια για ποια εγκλήματα θα διώκουν και βεβαίω πλήττεται και η νομική βεβαιότητα. Εγώ λοιπόν αυτή την ε, κριτική που ασκούν τα εθνικά κοινοβούλια θα την ε, συμφωνήσω και νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι πως αγνοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο το θέμα. Αδελφός Μπάτεν, από το EFT. Thank you. Uh, e Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να δημιουργήσει μια εισαγγελία με τεράστιες εξουσίες σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Βρετανική κυβέρνηση ήδη έχει αναγγείλει πως δεν θα αποτελέσει μέρος του συστήματος όμως. Θέλει να συμμετάσχει στα 357 μέτρα αστυνομική και δικαστική συνεργασία, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο επικίνδυνα όσον αφορά τι παραδοσιακέ μα ελευθερίε. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, η απόφαση της ε, κυβέρνησης ε, να μιλάμε μέρος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι και άχρηστη και ανηλικρινής. Η χρήση όλων των ευρωπαϊκών μέσων όπως το Ευρωπαϊκό Εντέλμα και των νέων όπως η Ευρωπαϊκή Εντολή έρευνα, ε, την καθιστά βεβαίως συμβολική. Παρά το ότι λοιπόν δεν θα υπάρχει άμεση αρμοδιότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει de facto εξουσία μέσω των νομικών αυτών μέσων. Προσπαθεί λοιπόν, ε, εφόσον ξέρει πως δεν θα το δεχτεί κανείς το Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση να φέρει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την πίσω πόρτα. Αλλά για να προστατευτούμε θα πρέπει νομίζω να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει αυτό ψηφίστε UKIP στις ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Μπονανίνη από τους μη Grazie. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο για το θέμα που εξετάζουμε και ευχαριστώ τον συνάδελφο Γιακολίνο για το έργο του καθώς και τους υπόλοιπους συσκευητές. Θέλω να δηλώσω ότι συμφωνώ απόλυτα για το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι μια πρόσθετη αξία για το τομέα δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας. Είμαι λοιπόν υπέρ του να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο στη διαδικασία. Ε, ο Νομίζω ότι δυστυχώς οι απάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν μεγάλο εμπόδιο για τη λειτουργία της Ευρωζώνης και επομένως πρέπει να επιμείνουμε για την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου θα συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη και η αντίδραση των, Ευρωπαϊκών, συγγνώμη, των Εθνικών Κοινοβουλίων μας έδειξε πόσο δύσκολη είναι ε, να πετυχεθεί η ομοφωνία στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βέβαια, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει επιπτώσεις, οι εξουσίες της θα έχουν επιπτώσεις ε, στα δικαιώματα των πολιτών. Επομένως, δεν θα πρέπει απλώς να σταματήσουμε στο να δώσουμε συμβουλές ε, στο Συμβούλιο, αλλά πρέπει να αναφερθούμε και στην αναγκαιότητα να διασφαλίσει και την, ε, προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων των ανθρώπων. Υπάρχει μία μπλε κάρτα από τον ε, κύριο Άλμπρεχτ. Αν είναι για προηγούμενο μιλητή δεν μπορούμε να πάμε προς τα πίσω. Αν θέλετε να απευθυνθείτε στον κύριο Μπονανίνη. Καλώς. Για την κυρία Κάρι ζήτησα εγώ μπλε κάρτα, μα το είχατε προσέξει νομίζω. Όχι, αν ε, το είχα δει θα σας είχα δώσει το λόγο. Γιατί καθυστερημένα έφτασε το ετοιμάσεις και τώρα έφυγε η κυρία Κάρι. Μικρόφωνο παρακαλώ. Uh, what I have heard... Αυτό που άκουσα πριν από αυτόν, ίσως θα μπορεί να μου απαντήσει ο κ. Μπενανίνη, είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία. Προφανώς δεν χρειάζεται βελτίωση. Αλλά εγώ αυτό που έχω ακούσει μέχρι τώρα από τους εισαγγελεί και είμαι μέλος των Πρασίνων που είναι υπέρ των πολιτικών ευθεριών και της επικουρικότητας, αλλά αυτό που άκουσα είναι ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη για καλύτερη συνεργασία όταν μιλάμε για την επιβολή του νόμου. Έτσι λοιπόν θα, θα ήθελα να μου πείτε Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν αν θέλετε και εσείς να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Όμω, ο κύριος Μπονανίνε δεν είναι σε θέση, ούτε επιτρέπεται να απαντήσει εκ μέρου ενό άλλου, μια άλλη συναδέλφου. Επομένω προχωρούμε με τους επόμενους ομιλητέ. Ο κύριος Βό έχει το λόγο. Ε, Σα ευχαριστώ. Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι μια καλή ιδέα. Όσο εισηγητής όμως για τη μεταρρύθμιση του Τζάστα, θα ήθελα να τονίσω πως ε, υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα που πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν πριν εγκρίνουμε και εφαρμόσουμε την πρόταση για τα δύο αυτά θεσμικά όργανα. Πρώτον, τι θα γίνει με τη μεταρρύθμιση της Eurojust από εδώ και μπρος για την περίπτωση που θα έχουμε ενισχυμένη συνεργασία και παρενθετικά εδώ πέρα θεωρώ πως η βάση της ενισχυμένης συνεργασίας ε, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αντίφαση. Δεύτερον, ποια επίδραση έχει η σύσταση της αγγελίας στον προϋπολογισμό της Eurojust και επιπλέον όλη αυτή η Όλες αυτές οι διαδικασίες στον τομέα του ποινικού δικαίου γύρουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν όσον αφορά το δικονομικό δικαίο σεβόμενοι πάντα τα εθνικά συστήματα, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και βεβαίω ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ο δομέ σε κάθε κράτο μέλο. Πρακτικά λοιπόν, εάν το εφαρμόσουμε όπω το έχουμε τώρα μπροστά μα, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. γιατί για ποια ε, ανεξαρτησία μιλάμε όταν θα έχουμε ένα όργανο το οποίο θα δράσει λογικά. Τι συμβαίνει με τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Επίσης, τι γίνεται όταν μπορεί να επιλέξει ο εισαγγελέας το δικαστήριο στο οποίο θα εκδικαστεί η υπόθεση από ό,τι φαίνεται. Νομίζω λοιπόν πως έχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ήμουν Υπουργό Δικαιοσύνη ε, την ε, εποχή που μπλοκαριστική συνθήκη τη Λισαβόνα και υποστήριξα το άρθρο 86 τη συνθήκη τη Λισαβόνα και φυσικά συνεχίζω να την υποστηρίζω με το σημερινό μου ρόλο σήμερα, τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό τον αιώνα εγκρίνει μια θετική θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα σταδιακό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Το πρώτο βήμα μια εισαγγελία που θα μπορεί να ασκεί δίωξη κατά της απάτης και να περασπίσει τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα πρέπει να είναι ικανή και να επιβάλλει τη δικαιοσύνη και να διώξει το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Αυτό απαιτεί καταρχήν να διαφοροποιήσουμε πολύ καλά ε, τις αρμοδιότητες της Eurojust και της OLAF από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεύτερον, να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της, να θεσπίσουμε πολύ καλά τα όρια μεταξύ Εθνικών Εισαγγελιών και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επίσης, θα πρέπει να ξεπεράσουμε και τις θεσμικές δυσκολίες. κάποια εθνικά κοινοβούλια παρουσίασαν κεντρική κάρτα. Κάποιες εθνικές κυβερνήσει ε, δεν αναλαμβάνουν δράση, είναι διστακτικέ. Ε, θα έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή ίσως ε, και με την διευρυμένη συνεργασία και επίση θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε τον ενεργό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υπερασπίσουμε την πρακτική δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία госпожо председател. Уважаеми колеги, подкрепям създаването на Европейска... Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ πάντοτε στήριξα την ιδέα αυτή για ένα πακέτο ευρωπαϊκό το οποίο θα αυξήσει την πίστη και την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα εξασφαλίσουμε μια ομοιόμορφη εφαρμογή και ισότιμη εφαρμογή του δικαίου ε, και του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να σας πω πως χώρες ε, ε, όπως η Βουλγαρία, όπου η εισαγγελία είναι ένας θεσμός που θεωρείται σε εθνικό επίπεδο διεφθαρμένος. Και σίγουρα αυτή τη στιγμή ε, οι πολιτικοί οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν κοινοί εγκληματίες στα αεροπλάνα και πυροβολούν σε αυτοκινητοδρόμους δεν επιπλήττονται. Αυτό που πιστεύω είναι πως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τελικά. Κατά τη γνώμη μου θα είναι μια εγγύηση για κυριότητα, για επαγγελματισμό και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα κάνουν να μας πιστέψουν περισσότερο οι Βούλγαροι πολίτες. ευχαριστώ Πρόεδρε επιτέλους κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος ε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χάρη στην νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χάρη στο έργο του συναδέλφου τον ε, ευχαριστώ τον κύριο Κολίνο, για το έργο του για τη καλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, θα διασφαλιστεί μόνο αν λειτουργεί ταχαίως και αν δεν λειτουργεί γραφειοκρατικά. Πρέπει να είναι ανεξάρτητη, πρέπει να ε, είναι επαγγελματικός ο τρόπος λειτουργίας της ε, και θα πρέπει οι έρευνες να προστατεύουν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ένα μέσο για να εγγυηθούμε και να αναπτύξουμε αυτό το χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας ε, που εκφράζεται στη συνθήκη και να σεβαστούμε τις τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Θέλουμε να ελέγξουμε και το διασυναριακό έγκλημα και φυσικά ε, η δράση του οργανωμένου κλίματος γίνεται εμφανής και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Απέναντι σε τέτοια αδικήματα ε, δεν ε, αρκούν οι νομοθεσίες σε εθνικό επίπεδο οι οργανισμοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν τις εξουσίες για να ασκήσουν δίωξη σε ποινικό επίπεδο. Επομένως, καλωσορίζουμε ένα τέτοιο μηχανισμό και φυσικά να μένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Σκούρια, κύριο Καρόνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής εισαγγελία θα αποτελούσε ένα πρώτο βήμα, ένα σημαντικό βήμα, αν ε, και δεν θα ήταν ολοκληρωτικό στο πλαίσιο μιας ε, πιο στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα τόσο λεπτό θέμα όπως είναι αυτό της ποινική δικαιοσύνη. Είναι σημαντικό γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινούσε συγκεκριμένη διαδικασία εναρμόνισης μεταξύ των διάφορων νομοθεσιών για να φτάσουμε σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Γιακολίνο στο ε, κοινό ε, ευρωπαϊκό χώρο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνη. και επίσης ε, θα καταπολεμούσαμε και το διασυνοριακό έγκλημα. Μπορούμε να πούμε ότι στα διάφορα εθνικά κράτη το έγκλημα πολύ γρήγορα έλαβε μια διάσταση πέραν των συνόρων. Επομένως, πέρα από τις ε, αντιδράσεις που είδαμε από τα κράτη-μέλη να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει και μια πολύ περιορισμένη δράση. Εγώ νομίζω λοιπόν σε αυτό το θέμα θα χρειαζόταν μεγαλύτερο θάρρος από δικής μας πλευράς για να δώσουμε κοινέ απαντήσεις σε κοινέ προκλήσεις. Ευχαριστώ κύριε Καρόνα. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το διασυνοριακό έγκλημα αυξάνεται στην Ευρώπη και πρέπει να αυξηθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να το καταπολεμήσουμε. Δεν θα πρέπει να μπορούν να κρυφτούν πουθενά οι εγκληματίες στην Ευρώπη. Η εντολή του Ευρωπαίου Εισαγγελία θα πρέπει να περιοριστεί στη βλάβη των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Και δικαίως Τίθεται όμω εδώ πέρα ένα ζήτημα για την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και Ένωση. και η προσθέμενη αξία εδώ πέρα είναι κάπω αμφίβολη. Η εισαγγελία μπαίνει στα εθνικά νομικά συστήματα σε τομεί του ποινικού δικαίου, όπω παραδείγματο χάρη το παραδεκτό των αποδεκτικών στοιχείων, προσφυγή κατά των αποφάσεων τη εισαγγελία. Η σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών αρχών και Ευρωπαϊκή εισαγγελία υπονομεύει την νομική βεβαιότητα η δομή δεν είναι σαφής. Τι θα γίνει στην πραγματικότητα με εθνικούς αντιπροσώπους, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα, θα συνεχίσουν οι έρευνες να γίνονται από ε, θα πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται οι έρευνες από εθνικούς εισαγγελείς για να μην υπονομευτεί η δικαιοσύνη. Επίσης θα πρέπει να οριστούν ξεκάθαροι οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφωθεί μια πρόταση που θα σέβεται καλύτερα την επικουρικότητα. 14 εθνικά κοινοβούλια που έβαλαν κίτρινη κάρτα δεν μπορούν να γνωριθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο. Πρέπει να σας πω πως η ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δημιουργηθεί για να διώκει το έγκλημα ε, και για να παραπέμπει στην δικαιοσύνη όσους καταπατούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω πως χρειαζόμαστε μια αποκεντρωμένη δομή η οποία θα πρέπει να βασίζεται στα όσα θεσπίζει το εθνικό δίκαιο των διαφόρων κρατών μελών. Γιατί ξέρετε πως τα αδικήματα είναι πολλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε παράνομες δραστηριότητες, ε, απάτη ΦΠΑ, διαφθορά, ε, ταμεία συνοχής, απάντηση σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα γεωργικά ταμεία, λαθρεμπόριο, λαθρεμπόριο τσιγάρων, οπότε υπάρχει πεδίο δόξας λαμπρό. Θα ήθελα να σχολιάσω πως χρειάζεται μια ξεκάθαρη ε, διάκριση αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών μεταξύ Eurojust, Europol ε, και εισαγγελία. Ο συνάδελφος Νίκολσον. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία που παρουσιάστηκε για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν η καταπολέμηση της απάτης ε, για την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και ορισμένα από τα ποσά ήταν εκπληκτικά πέρσι. Ε, μιλήσαμε για 104 εκατομμυρία που χάθηκαν λόγω απάτης ε, και από ό,τι φαίνεται μάλλον 12 φορές παραπάνω ήταν αυτό το νούμερο η Ευρωπαϊκή συγκυρία είναι ο καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε την απάτη. Νομίζω αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί. Στην ε, δική μου εκλογική περιφέρεια, ίσως ε, περισσότεροι νομίζουν ε, ότι τα θέματα της αστυνόμευσης είναι πάρα πολύ λεπτά και μετά από πολλά χρόνια αλλαγών η εμπιστοσύνη του κοινού στην αστυνόμευση στη Βόρεια Ιρλανδία οικοδομήθηκε. Εγώ είχα τότε κάποιες επιφυλάξεις και νομίζω τους τελευταίους μήνες είδαμε ότι ε, πόσο λεπτή μπορεί να είναι αυτή η εμπιστοσύνη. Και τα τελευταία νέα από τη δική μου εκλογική περιφέρεια ήταν ότι υπάρχουν κάποιε ανησυχίε που πρέπει να ακούσουμε. Μπορώ να πω ότι η προσέγγιση μηδενική ανοχή για την απάτη ε, στον προβληματισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη, αλλά αυτό αφορά ε, τώρα την δημιουργία της Νέα Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, εγώ θεωρώ ότι αυτή δεν είναι απαραίτητη λύση, γιατί είναι μια δαπανηρή λύση. Κάτσε διάει, πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και πρώτα θα παρακαλέσω τον συνάδελφο Στίερ. Ευχαριστώ, predsjednice, εγώ πρώτον prvom redu ρέτσι, τα da ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω πως στηρίζω αυτή την έκθεση και στηρίζω και αυτή την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το είπα ήδη από τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν είναι απλά φυσικό να έχει και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να υπερασπίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προστατεύει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Επίσης θα πρέπει να επεκταθεί ο χώρος του ποινικού δικαίου στην Ευρώπη. Αυτό που ζητάμε είναι να είναι ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τις εθνικές κυβερνήσεις, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να μην υπάρχει καθόλου πολιτική επιρροή. Επίσης θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Και ας πω εδώ πως η αρχή της επικουρικότητας δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για να κρύψουμε κάποια κάποιους τρόπους με τους οποίους ασκείται πολιτική πίεση και επιρροή στις εθνικές εισαγγελίες. Χαιρετίζω την έκθεση και καλώ όλα τα κράτη-μέλη και τους βουλευτές να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είμαι υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών, ειδικά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα και την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες. Αντί να φτιάξουμε όμως άλλον ένα φορέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι εθνικοί μηχανισμοί και η δικτύωσή τους. Θα είναι δύσκολο και επικίνδυνο να έχουμε μια κατάσταση όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία σε δύο επίπεδα γιατί έτσι θα υπάρχει σύγχυση και πρόβλημα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σκοπεύουμε να αποτελέσει η εισαγγελία μέρος των εθνικών δομών, αλλά έτσι θα δημιουργηθεί ένα προς το βάρος το οποίο δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Εγώ κατανοώ όλε τι ανησυχίε των προηγουμένων ομιλητών. Είπαν ότι δεν μπορεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τα χρηματοδομικά τη συμφέροντα. Πρέπει να σκεφτούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Για να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα και να το αναχαιτήσουμε. Δεν πιστεύω όμω ότι η δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο κατάλληλο τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι ως προς το συντονισμό των ε, δραστηριοτήτων ε, και να συντονίσουμε τις ε, εισαγγελίε των κρατών μελών. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε βελτικές πρακτικές, ανταλλαγή πληροφοριών, κατάρτιση και πιστεύω ότι η δημιουργία αυτής της εισαγγελία θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ διάφορων εισαγγελιών σχετικά με τις αρμοδιότητες ε, και τα όρια. Και εγώ νομίζω ότι θα υπάρχουν και μεγαλύτερες ε, δαπάνες. Ζούμε μια μεγάλη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να δαπάνουμε χρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι πως ε, φαίνεται να ακολουθεί κάποια λογική αυτή δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όντως, ενδεχομένως να γίνονται απάτες και να πλήττονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως αυτή η καλύτερη απόκριση, θα είναι αποτελεσματική η Γενική Εισαγγελία αυτή η Ευρωπαϊκή. Γιατί διαφορετικά μιλάμε για μια ε, απώλεια χρημάτων χωρίς να εξυπηρετείται κάποια από τα συμφέροντά μας. Ένα άλλο ερώτημα. Τι είδους δικαστήριο θα έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Θα έχουμε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο, θα έχουμε Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, γιατί δεν έχουμε λάβει ε, κάποια απάντηση στα θέματα αυτά. Αντίθετα, έχουμε 14 ε, εθνικά κοινοβούλια τα οποία έχουν σηκώσει κίτρινη κάρτα, ρεκόρ αριθμός ρεκόρ. Σας παρακαλώ να αποσύρετε ε, την πρότασή σας για να μην έχουμε επανάληψη των όσων έγινε στην ψηφοφορία σήμερα το πρωί όπου η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πλειοψηφία απορρίφθηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. i nadam se da će se na taj način postići stvarno prostor zajedniki prostor Λοιπόν, αυτό γίνεται διασυνοριακά. Μια τέτοιου είδου εισαγγελία θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε έναν ενιαίο χώρο δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Πρέπει να υπερασπιστούμε και να φροντίσουμε αυτά τα ε, συμφέροντα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Είναι κοινό ο στόχο τη πάταξη τη απάτη γιατί βεβαίως η απάτη υποσκάπτει την εμπιστοσύνη που δείχνουν προς εμάς οι πολίτες μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας κατευθύνουν οι διατάξεις οι οποίες ε, βρίσκονται στην ε, χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων, βεβαίω ε, θα πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Αλλά ίσω θα έπρεπε τα κονδύλια αυτά να πάνε κάπου αλλού. Επόμενο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα απλά να υπογραμμίσω πως ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βασίζεται στο άρθρο 86 της συνθήκης, συγκεκριμένο άρθρο το οποίο λέει, περιγράφει το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την ασυνήθιστη νομοθετική διαδικασία. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την επικοδομητική στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας και βεβαίω. Ε, αναμένα την ε, έγκριση της ενδιάμεσης έκθεσης. Συμφωνώ οπωσδήποτε με το Κοινοβούλιο πως δεν είναι δυνατόν να έχουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς δικαιώματα ε, του κατηγορουμένου τα οποία θα προστατεύονται με τρόπο οριζόντιο και βεβαίως ε, αντιλαμβάνομαι γιατί η Κομισιόν το υπογράμμισε αυτό και θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την στήριξή του για τα δικονομικά δικαιώματα και για το ότι ζητάει από το Συμβούλιο να εγκριθούν τα δικαιώματα αυτά τα οποία εκκρεμούν. Σας ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε και τώρα ο εισηγητής μας, ο κύριος Γιακολίνο. Ναι, Άκουσα φορές επικρίσεις, εκτιμήσεις ε, για ένα φάκελο, για ένα θέμα που ενδιαφέρει τα μάλα τους πολίτες. Ε, θέλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή μία αρχή που υπάρχει στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει ταυτόχρονα όμως να υπενθυμίσουμε σε όλους τους αδελφούς ότι πρόκειται για μια ενδιάμεση, για μια προκαταρκτική έκθεση και θέλαμε εδώ να αντιμετωπίσουμε κάποιες επικρίσεις απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν. Γενικά πάντως είμαστε θετικοί απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν, δικονομικά δικαιώματα, εγγυήσεις, να αξιολογήσουμε με ακρίβεια το κόστος, να έχουμε έναν ξεκάθαρο ορισμό για το φυσικό δικαστή, ε, να υπάρχει δέσμευση, ανάληψη των κατάλληλων εξουσιών από την Ευρωπαϊκή Συγγελία φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και μία αναθεώρηση της ε, Όλαφ ε, όταν θα τεθεί σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θέλουμε μία εισαγγελία που θα καταπολεμά ε, τις απάτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που θα λαμβάνει ταχύτατα αποφάσεις. Θα πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά και γρήγορα να προστατεύει τους πολίτες, να προστατεύει τα δικαιώματα του κατηγορούμενου και να διασφαλίζει ότι θα λαμβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις. Έτσι οι πολίτες θα μπορούν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στα ευρωπαϊκά όργανα, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διασφαλίσει ε, ε, πόροι που διαφορετικά όπως ε, ξέρετε θα φερούνταν για να χρησιμοποιηθούν ε, υπέρ εγκληματικών συστημάτων. Προτείνω λοιπόν να ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους υπενθυμίζοντας και την εργασία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και πιστεύω ότι και αύριο θα υπάρχει υποστήριξη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα κάνει ένα βήμα προς την έγκριση του τελικού κειμένου. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Η ζήτηση για την έκθεση του κυρίου Γιακολίνο ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία, όπως είπε και ο ίδιος, θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2013. Και θέλω πρώτα να παρακαλέσω εξ ονόματος του Συμβουλίου τον